Αύριο στις 10.30 θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή. Τέλος. Έχουμε μια σύντομη παρουσίαση της έκθεσης της κυρίας Μεγγέλης Ράμος για την εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό με τα φώτα που έγινε πριν ήταν υπέροχο. Πρέπει να το επαναλάβετε. Να γίνεται πιο συχνά εδώ στην Ολομέλεια. Κυρίως για μας που είμαστε εδώ στη νυχτερινή ήταν πραγματικά σαν να βλέπαμε το ξημέρωμα. Κύριε Πιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, για να διατηρήσουμε τα οικοσυστήματα και να λάβουμε υπόψη μας τα αλληλευτικά αποθέματα, να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, να βελτιώσουμε την γνώση όσον αφορά την τεχνολογία και την καινοτομία, είναι στόχοι που δεν μπορούν να επιτεθούν αν δεν έχουμε την στήριξη της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας. Η έρευνα στην Αλία επίσης είναι κάτι αναγκαίο για να καταλήξουμε σε συστάσεις και αξιολογήσεις που θα προτείνουμε στους νομοθέτες. Έρευνα για την ανάπτυξη έτσι όπως τα ξέρουμε σήμερα ε, μπορούν να βοηθήσουν ώστε να έχουμε μια καλύτερη κοινή ελευθερική πολιτική. Όμως ένας ε, επιστήμονας είπε κάποτε ότι το πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα, αλλά οι ανθρώπινοι πόροι. Η έρευνα στον τομέα της αηλίας ε, δεν είναι μόνο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι διτό, κύριε Επίτροπε. Γιατί από τη μια τα ποσά τα οποία γράφονται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για την έρευνα στην αηλία που θα πρέπει να είναι κάτι το εγκάρσιο, από ό,τι φαίνεται δεν φτάνουν για να αντιμετωπιστεί το θέμα της έρευνας στην Ελία. Έπειτα, οι επιστήμονες. Και να ξέρετε ότι έχω μιλήσει με πολλούς επιστήμονες πριν φτιάξω την έκθεσή μου αυτή και πριν την ξεκινήσω και κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της. Προβληματίζονται κάθε φορά που πρέπει να υποβάλουν προγράμματα για το εβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Και γιατί. Γιατί από τη μια έχουμε την, τις ηχθοκαλλιέργειες και από την άλλη μεριά έχουμε την έρευνα στους ωκεανούς που είναι ένα πολυκλαδικό ζήτημα. Στο έβδομο πρόγραμμα δράσης πάντως και τα δύο θέματα καλύπτονταν από τους ίδιους πόρους και εξαρτώνταν από την Γενική Διεύθυνση Αλίας. Τελικά το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους επιστήμονες για το πώς ε, να πείσουν τους υπαλλήλους για τις ανάγκες και τις ανησυχίες του τομέα. Έπειτα, η επιστημονική κοινότητα πιστεύει ότι η Γενική Διεύθυνση προτίμησε τη βασική έρευνα, χωρίς να δώσει τη σημασία που θα έπρεπε στην εφαρμοσμένη. Από πλευράς επιστημονικής, για παράδειγμα, η έρευνα στην Αλία που συνδυάζεται με το περιβάλλον. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θάλασσα θέλει ένα καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον και αλλιεύματα. Αυτά όμως απαιτούν επιστήμονες που δουλεύουν βάσει μιας οριζόντιας χρηματοδότησης στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Πάντως είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι επιστήμονες στον τομέα αυτό. Και γιατί, από ό,τι φαίνεται, επειδή η επαγγελματική ε, ζωή με τους τομείς αυτούς δεν φαίνεται αρκετά ελκυστική για τους νέους. Υπάρχουν άλλοι τομείς που δίνουν διεξόδους επαγγελματικές πιο εύκολα στους νέους. Όμως πρέπει να είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα κάθε φορά στην έρευνα, να έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα και για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Ινστιτούτων. Και αναγκαίο επίσης είναι να λάβουμε υπόψη μας και την εμπειρία των ίδιων των αλλιέων κάθε φορά που ετοιμάζονται επιστημονικές εκθέσεις βάσει των οποίων αποφασίζεται η ελευθερική μας πολιτική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε, κύριε Μιγκουέλες Ράμος. Το το Λόγω στον κύριο Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό να μιλάμε για την τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ευθύνης. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την, εφαρμοσμένη... την έκθεση για την εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της κοινή ε, ελευτικής πολιτικής και την εξαιρετική δουλειά της κυρίας ε, Μιγγέλες Ράμος. Η έκθεση αυτή έρχεται την κατάσταση κατάλληλη στιγμή και συνδυάζεται με το, την κατάρτιση του προγράμματος 2010 για το πρόγραμμα πλαίσιο 7 όπου αναφέρεται και η αλληλεία και η έρευνα και βασικά συμφωνούμε με τις ε, κεντρικές ιδέες της εκθέσεως ε, στηρίζουμε την ε, προσπάθεια διότι οι προτεραιότητες αυτές υπήρχαν για να αναλυφθούν διάφορες πρωτοβουλίες και να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις ε, θαλάσσιες και ναυτιλιακές προσπάθειες και τη συνεργασία στους χώρους αυτούς μεταξύ των κυβερνήσεων. Επίσης όσον αφορά την αλληλεία θέλουμε να την στηρίξουμε συγχρόνως όμως ισοσκελίζοντάς την με τους άλλους τομείς, τη δασοκομεία, τη γεωργία και ε, έχουμε ένα ε, ετήσιο προϋπολογισμό του προγράμματος πλαισίου 7 το οποίο βαθμιαία θα αναπτυχθεί και θα επωφεληθεί και ο χώρος αυτός από την αύξηση. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τονίσει περισσότερο την αλληλεία και τη γεωργία στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 και να στηρίξει και την έρευνα στους τομείς αυτούς, να στηρίξει τις κοινωνικές επιστήμες, και να ε, ζητήσει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει στην ε, ολοκλήρωση ε, της, της προσπαθίας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και φαντάζομαι ότι βάσει αυτών των πρωτοβουλειών έχουμε καλή βάση τώρα να βελτιώσουμε βελτιώσουμε και τη γεωργία και την αλληλεία με καινοτόμα έρευνα βάσει του νέου προγράμματός μας και να υποφεληθούμε από το συντονισμό της έρευνας μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλειών και των κοινών στόχων ε, της ελληνικής πολιτικής και πρέπει να σας πω ότι δεν είναι πιο περίπλοκο από ό,τι ήταν στο παρελθόν διότι ούτως ή άλλως οι ίδιοι άνθρωποι επεξεργάζονται τα ίδια θέματα και η συνεργασία που έχω με τον κύριο Μπόρτζ είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι αυτή, αυτό είναι το είδος ε, έρευνας που πρέπει να γίνεται διότι συνεργαζόμαστε καλά και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα τα οποία δεν θα είχαμε αν υπήρχε μεγαλύτερος κατακαιρματισμός μεταξύ των τομέων. Σας ευχαριστώ για την εργασία που κάνατε γιατί νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 10.30. Η επόμενη συνεδρίαση είναι αύριο 5η 19 Φεβρουαρίου στις 9 και επιτέλους μπορούμε να σβήσουμε τα φώτα και να λύσουμε τη συνεδρίαση. Καληνύχτα σας.